Καλημέρα. Συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση. Δύο ανακοινώσεις μετά τη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου που αναλάβαμε από τις πολιτικές ομάδες και από τους βουλευτές. Μία εγγεγραμμένη για για τους διορισμούς ε, με βάση το άρθρο 223. Οι κατάλογοι της σύνθεσης θα δημοσιευθούν στο site του Κοινοβουλίου και θα προσαρτηθούν στα πρακτικά. Μια άλλη ανακοίνωση. Το ΕΛΚ μου κοινοποίησε κάποιες αποφάσεις που τροποιούν τη σύνθεση των επιτροπών. Αυτές οι αποφάσεις θα υπάρχουν στα πρακτικά από τη σημερινή ημέρα. Με βάση τη μερίσια διάταξη θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Κομισιό, προετοιμάζοντα το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη 20 Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι παρούσα και χαιρετίζω την Υπουργό Μπρνάτ. Τη δίνω και το λόγο για την παρέμβασή τη. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, χαίρομαι πολύ που μπορώ να απευθυνθώ στην Ολομέλεια για να συζητήσουμε την προετοιμασία της ειδική ε, συνόδου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στις 20 Φεβρουαρίου. Μετά την παρουσίαση της Κομισιόν των προτάσεων για το επόμενο πολιετές η Βουλγαρική, Αυστριακή, Ρουμανική, Φιλανδική Προεδρία εργάστηκαν πολύ και σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο για να προλυάνουν το έδαφος για συμφωνία. Τώρα έχουν μπει σε μια αποφασιστική φάση μετά τη συζήτηση του Δεκεμβρίου κατά τη Σύνοδο. Το Συμβούλιο έκανε πολλές διαβουλεύσεις με τους ομολόγους. Επ' αυτής της βάσης θα υποβληθεί στις 17 Φεβρουαρίου προτάσεις στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, για συμφωνία. Η Κροατική Προεδρία υποστηρίζει την άποψη ότι η συμφωνία πρέπει να εξευρεθεί γρήγορα. Δεν θα είναι εύκολο, το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά εν πολλής ε, υπάρχει ε, κενό προσδοκιών μεταξύ αυτού που θέλουμε να πετύχουμε σε ενωσιακό επίπεδο και μεταξύ των κονδυλίων που χρειάζονται γι' αυτό. Όμως ε, η αναβολή δεν διευκολύνει τα πράγματα αντιθέτως. Το Brexit δημιουργεί δημοσιονομικό κενό το οποίο δυσκολεύει περισσότερο την κατάσταση ενώ η Ένωση ταυτόχρονα αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις και έτσι και προτεραιότητες. Μια ισορροπημένη συμφωνία που θα αντικατοπτρίζει φιλόδοξους στόχους της ε, στρατηγικής ατζέντα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Φεβρουάριο χρειάζεται για να ανοίξει ο δρόμος για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις επί πολλών εκκρεμών θεμάτων, ε, φακέλων συναπόφασης που πρέπει πρέπει να είναι έτοιμη για το νέο κύκλο τον Ιανουάριο του 2021. Χρειάζεται ο κανονισμός σε επίπεδο Συμβουλίου ε, να εγκριθεί γρήγορα. Αυτό δεν είναι άλλωστε το τέλος της υπόθεσης γιατί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συγκατατεθεί στο κανονισμό. Ε, γνωρίζομαι τη θετική συμβολή του, του, του Κοινοβουλίου. Ε, καθ' όλη την ε, πορεία ενημερώναμε το Κοινοβούλιο με τακτικές ε, συναντήσεις πριν και μετά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, συζητήσεις για το πολιετές και θα γίνει η επόμενη, την επόμενη εβδομάδα. Η Προεδρία μας θα συνεχίσει αυτή την πρακτική. Όποτε είναι στην επίσημη ημερήσια διάταξη το πολιετές. επίσης, το πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε πολλές υψηλού επίπεδου συναντήσεις με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου. Όταν βρεθεί ομοφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Κροατική Προεδρία θα εργαστεί σκληρά με το Κοινοβούλιο για ένα αίσιο αποτέλεσμα όταν θα ψηφιστεί από εσάς ο κανονισμός. Πρέπει έγκαιρα να βρεθεί ισορροπημένη συμφωνία για όλο το πακέτο του πολιετούς και του ιδίου πόρους. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων των θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των πολιτών. Ελπίζω ότι θα επιτύχουμε το στόχο μας αυτό. Η Κροατική Προεδρία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Πράγματι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το έκτατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είναι μια σημαντική στιγμή για την Ευρώπη γιατί η θέση εκκίνησης ε, η αφεντηρία είναι καλή, γιατί και τα τρία θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν συμφωνήσει για την ε, στρατηγική ημερήσια διάταξη. Και όλοι γνωρίζουμε περί τίνο πρόκειται εδώ. Έχουμε πολύ ξεκάθαρου κοινού πολιτικού στόχου. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι η πρώτη ουδέτερη προ το κλίμα Ήπειρο το 2050, όχι μόνο επειδή διακυβεύεται η υγεία των πολιτών. Αυτό είναι ο βασικό στόχο να την κατοχυρώσουμε την υγεία, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι αν έχουμε ένα καθαρό και φιλικό προς το περιβάλλον, ε, μια καθαρή και φιλική προ το περιβάλλον οικονομία, θα δημιουργηθούν βιώσιμε θέσεις απασχόλησης. Θέλουμε να αποφεληθούμε από την ψηφιακή αλλαγή στον κόσμο και θέλουμε να αναλάβουμε εδώ ενεργό ρόλο. Και θέλουμε να ενισχύσουμε τους πολίτες της Ευρώπης ε, με το να απο... πετύχουμε από τη μία τη μετάβαση μέσω τη οικολογική και ψηφιακής ε, μετάβαση, από την άλλη ε, επενδύοντα την εκπαίδευση ακριβώς ε, βάσει δεξιοτήτων στο ψηφιακό και οικολογικό τομέα. Ωστόσο δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί εάν ε, στο, δεν αποφασίσουμε τον προπολογισμό, το επόμενο έτος δεν θα είμαστε σε θέση να μπορέσουμε με τον νέο προπολογισμό, με τις νέες προτεραιότητες, πράγματι να μπορέσουμε να προβούμε στη χρηματοδότηση την οποία επιθυμούμε. Μετά από δύο χρόνια διαβουλεύσεων, ήρθε η ώρα να βρούμε κοινό έδαφος και πρέπει να βρούμε και τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις παλιές προτεραιότητες και στις νέες προτεραιότητες. Αν κοιτάξετε τις διαπραγματεύσεις, υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη τα οποία υπερασπίζονται στεναρά την πολιτική συνοχή και δικαίω. Υπάρχουν και πολλά κράτη-μέλη τα οποία υπερασπίζονται στεναρά την κοινή γεωργική πολιτική και δικαίω. Περιμένω όμως να δω την ίδια αφοσίωση για την υπεράσπιση των νέων προτεραιοτήτων. Γιατί τη μέρα που θα υπογραφεί ο προπολογισμό, αφού συμφωνήσουμε, όλοι θα στραφούν προς το Κοινοβούλιο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ζητήσουν τον ορίζοντα Ευρώπη, θα ζητήσουν το Εράσμο, θα ζητήσουν για ταμεία για τη μετανάστευση, για την άμυνα, για την ψηφιοποίηση, για τις υποδομές, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και επομένω, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι νέες προτεραιότητες εξασφαλίζουν την προσοχή που τους αξίζει. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός προπολογισμό, ο οποίος είναι σε θέση να μας δώσει την αυτότητα να επενδύσουμε σε νεοφύσει επιχείρησει, να εδραιώσουμε τη θέση της Ευρώπης ως ηγετικής δύναμης στην έρευνα, να δώσουμε δυνατότητες σε νέους, να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές κρίσεις μετανάστευσης να δείξουμε αλληλεγγύη σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών ή φυσικών κρίσεων και καταστροφών. Να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε ένα προϋπολογισμό ο οποίος για τους πολίτες και τις εταιρείες είναι ικανός να αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή. Για τους πολίτες αυτή είναι η ύψιστη προτεραιότητα. Για μας είναι μια πρόκληση. Είναι το καθήκον μας να κάνουμε αυτή την πρόκληση ευκαιρία. Και γι' αυτό, αγαπητοί βουλευτές, η επιτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό εξαρτώνται από τα μέσα που θα έχουμε για να χρηματοδοτήσουμε την πράσινη συμφωνία, τον Green Deal δηλαδή για την Ευρώπη. Δεν θα δεχτώ κανένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα εξασφαλίζει τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού να δοθεί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Περιμένω επίσης ένα προϋπολογισμό ο οποίο θα δίνει νέους πόρους, απαραίτητου πόρου, στον μηχανισμό για μια δίκαιη μετάβαση. Ο λόγος είναι απλός. Εάν δεν έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να στηρίξουμε τις περιφέρειες και τους εργαζόμενους, του πιο εκτεθειμένους στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, δεν θα καταφέρουμε απλούστατα να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα. Η Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη θα γίνει μαζί με τους πολίτες της Ευρώπης, μαζί με τους Ευρωπαίους ερευνητές, μαζί με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ή απλώς δεν θα γίνει καθόλου. Δεν θα υλοποιηθεί καθόλου. Και πιστεύω, όπως και εσείς, ότι νέοι ήδη για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μια σημαντική πρόοδος. Ακριβώς γι' αυτό Ζήτησα επιτακτικά από τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Είμαι πεπισμένη ότι έτσι θα επιταχύνουμε το κοινό μας πρόγραμμα και θα ελαφρύνουμε την πίεση που ασκείται στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν οι επιπλέον πόροι είναι μια λύση κερδοφόρα από κάθε άποψη. Αγαπητοί βουλευτές, ξέρουμε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες. Ως Ένωση των 27, όπως είπατε, θα έχουμε λιγότερους πόρους. 75 δισεκατομμύρια λιγότερα για την 7 ετία. Αλλά περισσότερες κοινέ προκλήσεις που κανένα κρατός μάλλον δεν μπορεί να επιλύσει από μόνο του. Παράλληλα, οι προσδοκίες για τον επόμενο μακροχρόνιο προπολογισμό της Ένωσης είναι πολυπίκυλε ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις συζητήσεις που γίνονται στις δικές σας χώρες και βλέπετε και τις διαφορετικές θέσεις στα κράτη-μέλη των συναδέλφων σας. Το να φτάσουμε σε συμφωνία θα είναι μια δύσκολη υπόθεση. Το ξέρουμε, θα είναι μια πρόκληση. Αλλά ξέρουμε επίσης ότι οι πολίτες δεν θα καταλάβουν αν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν μπορέσουν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για τις πολιτικές που είναι απαραίτητε. Είναι κοινή μας ευθύνη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα καταφέρουμε για το καλό της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και τώρα θα ακούσουμε την άποψη των πολιτικών ομάδων. Ο Πρόεδρος Βέμπερ θα μιλήσει εξ ονόματος του ΕΛΚΑ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ε, συνάδελφοι, όταν μιλάμε για τον προπολογισμό, μιλούμε για την πολιτική, για το μέλλον της Ευρώπης. Πού μπορούμε να δώσουμε τις προτεραιότητες. Θα ήθελα καταρχήν να τονίσω ότι από, κατά την άποψή μας θα ήταν καλό να ήταν εδώ ο Σαλ Μισελ το να ακούσει τα όσα λέμε θα ήταν καλό. Γνωρίζουμε ότι έχει μια στενή, βρίσκεται στενή ανταλλαγή με του ειδικού μα, με το steering group, αλλά θα είχε μια άλλη βαρύτητα αν ερχόταν στην Ολομέλεια. Γι' αυτό θέλουμε να πούμε ευθύ εξ αρχή ότι θα ήταν καλό εάν βρισκόταν εδώ. Αλλά είναι θετικό το γεγονό ότι έθεσε την ημερομηνία ε, της 20 Φεβρουαρίου ε, πιέζει την Επιτροπή, προσπαθεί να δώσει απαντήσεις και ασφάλεια για τους πολίτες, για τους ε, γεωργούς, τους ερευνητές, τους φοιτητές. Όλοι θέλουν μια σαφήνεια εν σχέση με το μέλλον. Γι' αυτό το ευχόμαστε καλή επιτυχία για τις 20 Φεβρουαρίου. Έχουμε μια νέα εντολή, είναι κατάλληλη συγκυρία. Η Επιτροπή έχει επίσης μια φρέσκια εντολή. Όλοι έχουμε μια νέα ορμή και γνωρίζουμε τι θέλουμε για τη νέα και θα πρέπει να ορίσουμε τι θέλουμε για τη νέα Ευρώπη. Το πρώτο σημείο είναι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζητούμενο δεν είναι να υπερασπιστούμε τα εφιστάμενα μέσα κονδύλια. Ε, δεχόμαστε κριτική ε, και θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε και μία αυτοκριτική κατά πόσο έχουν τα ταπανηθεί σωστά τα κονδύλια. Ο Ιωάννης Χάνες ανέλαβε μία ευθύνη με τις προτάσεις, ως προς τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί, δηλαδή να ασκήσει μία αυτοκριτική. Αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά τον έλεγχο του προπολογισμού του, ώστε να τεθούν τα όρια για κάποιε πληρωμέ προ μεμονωμένα άτομα. Αν κάποια άτομα ε, λαμβάνουν τεράστια ποσά από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν μπορεί να είναι ορθό. Γιατί μιλούμε για ένα είδο αντιολιγαρχικού νόμου στην Ευρώπη, να μην καταλήγουν τα χρήματα σε λίγα χέρια. Δεύτερον, θα πρέπει να υπερασπιστούμε τις ε, υφιστάμενες ε, επενδύσεις. Οι γεωργοί χρειάζονται υποστήριξη, η ύπεθρος χρειάζεται υποστήριξη στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, η περιφερειακή ανάπτυξη ούτω ώστε να αυξηθεί η συνοχή της Ευρώπης και οι τομείς της έρευνας του Εράσμους ε, δείχνουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Το τρίτο σημείο που είναι σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε οικονομία όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Η γεωργία, η περιφερειακή ανάπτυξη, αυτά τα έχουμε τονίσει. Αλλά δεν είναι δυνατόν να δημιουργεί μια δυναμική η οποία ε, κάνει περικοπές στους μελλοντικού τομείς, τομείς του μέλλοντος της Ευρώπης. Δεν θα ήθελα να γίνει η συζήτηση του 1% ε, για το ανώτατο όριο. Αλλά να μιλήσουμε συγκεκριμένα για περιεχόμενα. Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει 10.000 ε, εμπειρογνώμονες να απασχολήσει, οι οποίοι να μπορούν, στη Frontex που να μπορούν να ε, επερασπιστούν τα σύνορά μας. Είναι απαράδεκτο να περικόπτεται από τη Φιλανδική Προεδρία κατά εν τρίτο αυτός ο προπολογισμό. Το ίδιο ισχύει και για την έρευνα. Για παράδειγμα, ε, η καταπολέμηση του καρκίνου ε, χρειαζόμαστε τα αναγκαία κονδύλια για να έχουμε επιτυχία. Και ε, στο Εράσμος ήδη έχω αναφερθεί και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιωχάνες και την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν για την ε, σαφήνεια, το ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα πρέπει να μπουν στην άκρη αυτή οι σημαντικοί τομείς. Ε, επίσης το ζήτημα των καθαρών πληρωτών. Εάν θέλουμε να έχουμε σωστά σύνορα στην Ευρώπη, να έχουμε ένα Marshall σχέδιο για την Αφρική, δεν πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα που πάνε πίσω στη Γερμανία, στις κάτω χώρες κλπ. Ε, ή στην Αυστρία. Α σταματήσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση για τους καθαρούς πληρωτές. Η, ε, η σωστή προσέγγιση είναι να δημιουργήσουμε τους ίδιους πόρους ε, και να πετύχουμε χρηματοδότηση με τους ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί πρόκειται για το κοινό συμφέρον των Ευρωπαίων, το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτείται με τους ευρωπαϊκούς ιδιού πόρους. Και θα ήθελα να πω, το Συμβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει ότι το ΕΛΚ όσον αφορά τους ιδίου πόρους, εδώ έχουμε μια κόκκινη γραμμή, γιατί χρειαζόμαστε μια συστημική αλλαγή της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα το τονίσουμε και στι διαπραγματεύσει για την προσχώρηση άλλων ε, χωρών. Επίση, το rule of law, το κράτος δικαίου, τα χρήματα της Ευρώπης ε, μπορούν να χορηγηθούν μόνο εφόσον τηρούνται βασικές ε, αρχές, η δικαιοσύνη, το θέμα των μέσων μαζική ενημέρωση κλπ. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ένας του κράτου δικαίου με το πολιτέ. Ο David Κάμερον στη τελευταία συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είπε ότι μόνο ένα, ε, θα πρέπει να είναι μόνο 1%, 1%, 1%, γιατί έτσι θα πείσουμε τους Βρετανούς ότι η Ευρώπη είναι αποτελεσματική και ε, στρέφεται προς το μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζήσαμε το Brexit. Εάν δώσουμε τροφή στους δημαγωγούς, στους λαϊκιστές, θα τους ενισχύσουμε και δεν θα τους αποδυναμώσουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Όχι τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή, αλλά μακρόπνοες ε, φιλοδοξίες για την Ευρώπη. Η πρόεδρος Γκαρσία Πέρεθ εκ μέρους των σοσιαλιστών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε ε, εν μέσω μιας συζήτησης πολύ σημαντικής που θα ε, σημαδέψει όλη την ευρωπαϊκή θητεία αλλά και το μέλλον της Ευρώπης. Ε, δεν αρκεί να θέσουμε τους στόχους εάν μείνουμε με δεμένα χέρια. Βρισκόμαστε σε μια σημαντική συγκυρία για την Ευρώπη, το γνωρίζουμε όλοι. Επίσης το Συμβούλιο το γνωρίζει. Γνωρίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται πραγματικά να, να κάνει μια, ε, ένα μετασχηματισμό για να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα στον κόσμο, ένα μετασχηματισμό στον οικονομικό, κοινωνικό, ε, τομέα ε, και στο περιβαλλοντικό. Το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζει και το Συμβούλιο. Αυτό το οποίο μας χρειάζεται είναι να μπορέσουμε να βάλουμε πάνω στο τραπέζι τα, τους αναγκαίους πόρους, τα αναγκαία μέσα για να προχωρήσουμε. Η πρόταση αυτού του Κοινοβουλίου είναι πολύ λογική και αντιμετωπίζει ακριβώς αυτή την ε, αναγκαιότητα. 1,3% του ΑΕΠ και επιπρόσθετη πόρη για τις νέες πολιτικές που πρέπει να προωθηθούν προκειμένου να προσεγγίσουμε τη σωστή μετάβαση σε αυτό το τομέα. Η πρόταση αυτού του Κοινοβουλίου είναι πολύ ξεκάθαρη και έχει μια μεγάλη πλειοψηφία στήριξη εκ μέρους των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Η πρόεδρος κυρία Βοντερ Λάιν επέμεινε στην ανάγκη να, έχουμε μια επιτροπή γεωστρατηγική. Και επίσης ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κ. Αλμισελ, Επίσης ανέφερε την ανάγκη να αγηθούμε τις μάχες για την κλιματική ευρωτερότητα στον κόσμο. Τώρα μας χρειάζεται να πείσουμε τους εταίρους μας στο Συμβούλιο. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή ότι θα θέλαμε και εμείς, ο κύριος Σαρλ Μισελ, να βρισκόταν εδώ. Ίσως ε, να έχει λίγα να πει, αλλά έχει πολλά να ακούσει. Και για να πείσουμε τους εταίρους μας στο Συμβούλιο είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε το μέγεθος ευθύνης μας και είναι αναγκαίο να έχουμε μπροστά μας μια συμφωνία που να μην υπάρχουν οι τιμένοι και οι νικητές γιατί με τρόπο αυτό αυτοί που θα χάσταν η Ευρώπη. Ε, το ζήτημα δεν είναι να πάρουμε χρήματα από τη μια πολιτική για να το πάμε στην άλλη ή χρήματα από μια περιοχή για να τα πάμε στην άλλη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ένα πράγμα. Ο Ζακ Τελόρ ήταν αυτό ο οποίο έθεσε εκείνη στο πρώτο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και έλαβε υπόψη ότι ήταν αναγκαίο να γίνει μια σημαντική ημερήσια διάταξη σχέση με την Ευρώπη πέραν των εθνικών συμφερόντων και ότι ήταν σημαντικό να προχωρήσουμε στην αλληλεγγύη του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Και αυτή είναι η φιλοδοξία που πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή. Ζητώ από τις επικεφαλείς των κυβερνήσεων ένα ευρωπαϊκό όραμα, γιατί βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή και αυτή τη στιγμή διακυβεύεται το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι είναι αναγκαίο να προσεγγίσουμε ε, δια, μια και καλή τους ιδίους πόρου με τα επιπρόσθετα κονδύλια τα οποία χρειαζόμαστε. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο προπολογισμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερου πόρου. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ για του νέου. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ για τον πρωτογενή τομέα, για του γεωργού και του κτηνοτρόφου. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική για να στηρίξουμε τους νέους επιχειρηματίες, τους ερευνητές κλπ. Είναι τόσο πολλές οι πολιτικές που χρειάζεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ε, που δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τη μάχη. Το ρολόι τρέχει και για μας μπορούμε να πούμε ε, ε, το εξή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει ισότιμα για τους όρους μαζί με το Συμβούλιο. Δεν πρόκειται να ενδώσουμε στην πίεση του χρόνου, γιατί το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στα χέρια μας και είναι η πιο σημαντική ευθύνη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Τζόρλος, εκ μέρους της ομάδας Renew Europe. Πρόεδρε, συνάδελφοι, η Ευρώπη αναμένεται να δώσει απαντήσεις στην μεταναστευτική κρίση, την κλιματοπιστωτική κρίση, την κλιματική κρίση, η μία κρίση μετά την άλλη πλήτη, την Ευρώπη. Περισσότερο παρά ποτέ η Ευρώπη είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητο να προσαρμόσουμε λοιπόν τον προπολογισμό σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Θέλω να χαιρετήσω την αποφασιστικότητα του Σαν Μισελ, που μαζί με την Κροατική Προεδρία προσπαθούν να βρουν συμφωνία πάνω στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τον στηρίζουμε πλήρω για να τα καταφέρει, αλλά υπό τον όρο ότι ο προπολογισμό θα είναι καλό προπολογισμό. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο μια υπόθεση δέσμευση. Παίρνουμε πολλέ πολιτικέ δεσμεύσει. Αναλαμβάνουμε πολλέ πολιτικέ δεσμεύσει τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε και εγγυήσει ότι αυτέ οι δεσμεύσει θα οδηγήσουν σε αυτά αποτελέσματα για τους προϋπολογισμούς. Και ένας καλός προϋπολογισμός δείχνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να δράσουμε μαζί. Και μόνο όταν έχουμε κοινέ πολιτικές φιλοδοξίες, θα είμαστε, με ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, θα είμαστε αξιόπιστοι. Οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής είναι απτές και πρέπει να δοθεί λύση, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Είναι απαραίτητο. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχή. Όλα αυτά απαιτούν Γρήγορε δράσει από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να τονίσω τρία πράγματα για την ομάδα μου. Καταρχά το μέγεθο του προπολογισμού. Χρειαζόμαστε τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει. Τα, με, τα τωρινά και τα μελλοντικά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μελλοντικέ καλέ φιλοδοξίε και να περιορίζουμε εμεί οι ίδιοι τι δυνατότητέ μα για να φτάσουμε σε αυτέ τι φιλοδοξίε. Είναι θέμα αξιοπιστία τη Ένωση απέναντι στου πολίτε. Οι πολιτικέ μα δηλώσει θα πρέπει να οδηγήσουν σε δράση. Ε, νέοι ή διπόροι, δεύτερον. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε αυτό το κομμάτι του προπολογισμού και να συνάδει με τι ε, συνθήκε. Ένα πραγματικό ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό σημαίνει στεναρή διποροι Η τελευταία μεταρρύθμιση του προπολογισμού έγινε το 1988. Είναι και η ώρα να εξυγχρονίσουμε αυτόν τον προπολογισμό. Τρίτον, ένα μηχανισμό ε, βασικός για το κράτος ε, δικαίου. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τον προπολογισμό όταν, προστατε... όταν γίνεται επίθεση στις αξίες της ε, Ευρώπης και το κράτο δικαίου. Ο... Το έρασμος, η απασχόληση για τους νέους, προστασία των συνόρων, άμυνα, διαχείριση της μετανάστευσης, όλα αυτά απαιτούν ένα καλό προπολογισμό μετά το Brexit, μετά τις κρίσεις που ζήσαμε συμφωνούμε ότι πρέπει να ανανεώσουμε την Ευρώπη. Η απόφαση για τον προπολογισμό θα πρέπει να είναι η απόδειξη ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δεχτεί ένα συμβιβασμό που υποσκάπτει την αξιοπιστία μια Ευρώπη ικανή να δρά προ όφελο των πολιτών τη. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο Τζάνι από την ομάδα ID. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Είναι κρίμα που ο πρόεδρος ε, Μισελ Σαρ Μισελ δεν είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Γιατί νομίζω ότι συγκαλέσαμε αυτή την έκτακτη σύνοδο και ήταν θέμα ε, αξιοπιστίας του ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Περιμένουμε τη νέα πρόταση για να δούμε τα νούμερα, για να δούμε αν άλλαξε κάτι, αλλά από τα νέα που μας έρχονται και από τις διμερείς επαφές δεν ε, φαίνεται ότι αυτή η πρόταση αποκλίνει πολύ από αυτά που είχε παρουσιάσει η Φιλανδική Προεδρία, που δεν άρεσε ούτε στα κρατημέλη, στο Συμβούλιο, ούτε στο Κοινοβούλιο. Είχε δυσαρεστήσει δηλαδή τους πάντες και την Κομισιόν επίσης. Λίγους μήνες μας χωρίζουν από την τελική προθεσμία για την εξέβρεση συμφωνίας για το Πουδουπού. Πρέπει να κλείσει η ονειροφαντασία και να είμαστε πιο ρεαλιστικοί να δεχτούμε ότι είναι περιορισμένοι οι πόροι. Είναι περιορισμένοι οι πόροι και συμφωνώ εδώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος από το ΕΛΚ. Γιατί, Γιατί συχνά αυτό το κοινοβούλιο δεν ήταν σε θέση πολλές φορές να αποφασίσει θετικά για τον προϋπολογισμό, να επιλύσει προβλήματα απατών. Για πολιτικούς λόγους συχνά δεν είχαμε θετικά αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι αυτό οδηγεί σε μία στάση των κρατών μελών που είναι πιο συντηρητική. Αν εμείς δεν μπορούμε να αποδείξουμε την ε, προστιθέμενη αξία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ε, προφανώς τα κράτη-μέλη διστάζουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει οδηγίες, ε, κανονισμούς, ψηφίσματα που ζητούσε πειθαρχία από τα κράτη-μέλη για τον προπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πειθαρχία στη διαχείριση του δικού μα προπολογισμού και στη διαχείριση των δικών μα πόρων. Πιστεύω ότι οι προτεραιότητε που υπάρχουν, οι βασικέ προτεραιότητε, αυτέ που είναι εγγεγραμμένε σε ευρωπαϊκέ συνθήκε, μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρί να ζητήσουμε επιπλέον πόρου. Η γεωργία, η αλεία, η στήριξη τη περιφερειακή ανάπτυξη, η πολιτική συνοχή. Νομίζω ότι υπάρχει χώρο σε αυτόν τον προπολογισμό για να χρηματοδοτήσουμε αυτέ τι προτεραιότητε χωρί να ζητήσουμε επιπλέον πόρου. Μπορούμε να κόψουμε τα 20 δισεκατομμύρια ε, Ευρώπη για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν να κάνουν με τις επιλογές των κρατών μελών. Μπορούμε να κόψουμε τα 13 δισεκατομμύρια για τα διάφορα ταμεία, ιδίω ας πούμε για την Τουρκία. Τέλος πάντων, το βασικό είναι να κάνουμε μια ρεαλιστική πρόταση και να βρεθεί μια συμφωνία των συντομότερων δυνατών. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να έχουμε ρεαλισμό και να σταματήσουμε τι όνειροφαντασίε. Δεν έχει νόημα να ονειρευόμαστε. Ο πρόεδρο Λαμπέρ έχει το λόγο εξ ονόματο των πράσινων. Πιτή συνάδελφοι, ο προπολογισμό είναι ένα εργαλείο και γνωρίζετε ότι μπορούμε να συζητούμε για το μέγεθος του εργαλείου. Ε, το εργαλείο, ένα μεγάλο σφυρί, ένα μικρό σφυρί, παραμένει σφυρί. Ε, αυτό το οποίο θέλω να πω με αυτό είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Μου άρεσαν αυτά που είπατε κυρία Πρόεδρε, εκτός από το σημείο που είπατε ότι δεν θα δεχτώ ένα προϋπολογισμό όπου λιγότερα από 25% θα αφαιρεθούν στην κλιματική αλλαγή. Ε, και ε, βεβαίως εάν ε, τα υπόλοιπα ποσοστά αφιερώνονται τελικά στην επιδείνωση του κλίματος θα στοχίσουμε εντελώς. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή του συνολικού ευρωπαϊκού προπολογισμού σε σχέση με την οικολογική μετάβαση. Όσον αφορά την ΚΚΑΠ, δεν συμφωνώ γιατί ο στόχος της γεωρικής πολιτικής δεν είναι οι μεγάλες business αλλά να βοηθήσουμε τους ε, γεωργούς μας ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης προς μια οικολογική γεωργία. Όλα θα πρέπει να κατείνουν προς αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν το ζήτημα της ενοχής είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο θα μας επιτρέψει να κρίνουμε την ποιότητα της πρότασης του Συμβουλίου. Ε, ε, και δεύτερο στοιχείο, όπως είπε ο Μάνφρετ, η σύνδεση μεταξύ προπολογισμού και σεβασμού των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση αξιών πρωτίστως και όχι οικονομική. Και δεν μπορούμε να αποφεληθούμε από τα οικονομικά ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν παίζουμε με τους κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή σεβόμενοι τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πραγματικά δεν το έχουμε καταφέρει. Και βεβαίως ο όγκος είναι μια είναι ένα ζήτημα. 1,3% του ΑΕΠ είναι λογικό. Όλοι γνωρίζουν ότι μακροοικονομικά ε, ε, το, η μέγιστη επένδυση θα πρέπει να είναι το Green Deal. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τον πιλωτικό ρόλο που θα πρέπει να παίξουν οι δημόσιες επενδύσεις όσον αφορά τις υποδομές, στους σιδηροδρόμους για παράδειγμα. Εδώ χρειαζόμαστε ένα προϋπολογισμό αρκετά πλούσιο για να κάνουμε αυτές τις επενδύσεις. Ή, ή υπογράψτε για ένα ακόμα 3% ή να μου δώσετε τους ίδιους πόρους. Ε, κάνει το ίδιο, η σημασία είναι να προβούμε σε αυτή την αλλαγή. Και τελευταίο σημείο. Ε, ήμουν εδώ πριν από 7 χρόνια, την εποχή του Ζόζεφ Ντάλ, του Μάρτιν Σούλτς, του Φέρχοφ ε, Στάστ, ε, που έλεγαν πάνω από το νεκρό μας σώμα. Ε, δεν θα δεχτούμε αυτόν τον προπολογισμό γιατί σημαδοδεί μια πιστοχώρηση. Τι έγινε τελικά. Οι τρεις πρώτοι αποδέχτηκαν τελικά αυτό που είχαν ε, κρίνει ως απαράδεκτο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και εάν η πρόταση που θα υποβάλει το Συμβούλιο δεν ε, συνάδει με τους δικούς μας στόχους, δεν θα πρέπει να φοβε, φοβηθούμε τη σύγκρουση. Εμείς ε, δεν είμαστε ένα σώμα όπου απλώς ε, καταχωρούμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου και ο κύριος Μισελ έπρεπε να παρίσταται εδώ για να το ακούσει. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες που μίλησαν για το ότι θα έπρεπε ο πρόεδρο Μισελ να είναι παρόν, ούτω ώστε να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, λέει ο κύριο Φίτο, για το θέμα αυτό. Δεν θέλω να κάνω μια παρέμβαση παραθέτοντας τις προτεραιότητες. Πώς, μπορώ να μην συμφωνήσω με τις περισσότερους στόχους που αναφέρθηκαν. Δεν γίνεται. Οι ομιλίε που ακούμε μιλούν για την καταπολέμηση, α πούμε, της κλιματικής αλλαγής. Ποιος δεν συμφωνεί με αυτό θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το πώ θα την καταπολεμήσουμε. Μία παρέμβαση για την αύξηση τη καινοτομία, αύξηση των πόρων για του νέου, για του ερευνητέ. Και εγώ μπορώ να συμφωνήσω με αυτά. Μπορώ να συμφωνήσω με αυτέ τι απαριθμίσει προτεραιοτήτων που σχεδιάζουν μια πιο όμορφη και πιο καλή Ευρώπη. Το θέμα είναι όταν φτάνει ο κόμπο στο χτένι. Ποιοι είναι αυτοί οι κόμποι. Όταν πρέπει να κάνουμε λογαριασμού στον προπολογισμό. Και όταν έχουμε κινδύνους άμεσους απέναντι σε κάποια κράτη σε αντιδιαστολή με κάποια άλλα. Έτσι. Εκεί γίνεται η συζήτηση και εκεί μπερδεύεται το πράγμα. Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πολλές από τις πολιτικές, τις οποίες ακούσαμε να, αναφέρονται, να αναφέρεται η Επιτροπή. Θα πρέπει όμως για να τις εξασφαλίσουμε να περικόψουμε κάποιες γραμμές προϋπολογισμού που για το Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντική. Παραδείγματο χάρη πολιτική συνοχή και η κοινή γεωργική πολιτική. Λείπει το κουράγιο. Και το είπε κάποιο συνάδελφο. Και εγώ συμφωνώ με αυτό. Να κοιτάξουμε την αποτελεσματικότητα του προηγούμενου προπολογισμού. Δεν κάνουμε αποφασιστικές περικοπές σε κάποιες γραμμές προϋπολογισμού που δεν έδωσαν τα αποτελέσματα που θέλαμε. Δεν υπάρχει μια σαφής ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και να εξισορροπήσουμε τους, τις επενδύσεις για αυτό το θέμα. Η συζήτηση που ε, ξεκίνησε τη Δευτέρα για το Σύμφωνο Σταθερότητας ε, θα πρέπει να δείξει, ε, να μας δείξει κάποιο δρόμο. Ακούστηκε πάλι και σήμερα το πρωί το, θέμα του κράτους δικαίου. Έχουμε εδώ πέρα τον θεματοφύλακα των ευρωπαϊκών αξιών. Επομένως, πρέπει να μπορούμε να εξηγούμε τα κριτήρια που διέπουν το κράτος δικαίου. Πρέπει να μας εξηγήσει αυτός ο θεματοφύλακας. Και σε αυτή την περίπτωση, αν κάποιος δεν τηρεί το κράτος δικαίου, θα πρέπει να μην μπορεί να χρησιμοποιεί τους πόρους του προϋπολογισμού. Όλοι όσοι είναι εδώ μιλούν γιατί έχουν μια ε, νομιμότητα που τους δίνει η λαϊκή εντολή. Ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ ο κ. Παπαδημούλης. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η απουσία του Σαρλ Μισελ από τη σημερινή συζήτηση είναι απαράδεκτη και είναι και κακό σημάδι για όσα θα ακολουθήσουν. Κυρία Φόντερ Λάιεν, παρουσιάσατε ένα πρόγραμμα πενταετίας και πήρατε ψήφο εμπιστοσύνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό δεν είναι σωστό αυτό που λέει ο κύριος Χάν που κάθεται δίπλα σας ότι απλώς εσείς είσαστε ένας honest broker στη συζήτηση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Γιατί για να χρηματοδοτηθεί, το πρόγραμμα που εσείς παρουσιάσατε, χρειάζεται τουλάχιστον το 1,3 του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ που ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια τεράστια πλειοψηφία. Γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το Green Deal χωρίς να περικοπούν δραστικά οι πολιτικές συνοχής ή της κοινή αγροτικής πολιτικής και δεν θα υπάρχουν λεφτά για την καινοτομία για τις επενδύσεις και πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την επιβράδυνση της οικονομίας της ευρωπαϊκής αλλά και την πιθανή κρίση που έρχεται και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με έναν πιο φιλόδοξο προπολογισμό. και επειδή πρέπει να μιλάμε πρακτικά για να πετύχουμε έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό οι τρεις συνομοθέτες αυτός μπορεί να αναζητηθεί προς την πλευρά αυτών που προτείνει το κοινοβούλιο πάνω από αυτά που προτείνει η κομισιόν τα οποία είναι πια ξεπερασμένα κυρία φοντερ λάιεν γιατί ο προϋπολογισμός που παρουσίασε η κομισιόν ένα χρόνο πριν ως πρόταση είναι 5% κάτω από το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο. Και για να έχουμε αποτέλεσμα πρέπει κύριε Βέμπερ εσείς αυτά που είπατε εδώ να καταφέρετε να πείστε την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Κούρτς. Εσεί, κύριε Τσιόλο, αυτά που είπατε εδώ να καταφέρετε να πείσετε τον κύριο ρούτε και εσείς αγαπητοί ράτσε να πείσετε τους Πρωθυπουργού της δανίας και της σουηδίας. αλλιώς θα αναγκαστεί το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να ψηφίσει ένα προϋπολογισμό απαράδεκτο και αυτό κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει και δεν πρόκειται να συμβεί. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Πεντιτσίνη, εκ των μη εγγεγραμμένων. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή η πρόταση που είναι πιο κοντά στο δικό μας στόχο για το πολιτεύτημο συνομικό πλαίσιο είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προφανώς είμαι υπέρ. Και το είπαν και οι προλαλήσαντες προφανώς συμφωνούμε να στηρίξουμε σαφώς την Πράσινη Συμφωνία, τον Green Deal και τις πολιτικές που έχουν στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ε, κοινοτομίας. Πώς θα μπορούσαμε να είμαστε αντίθετοι. Πιστεύουμε επίσης ότι η καταπολέμηση της ε, μετανάστευσης θα πρέπει να στηριχθεί. Όπως και τα κράτη-μέλη που προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση αλλά αντιμετωπίζοντας και τις βαθιές αιτίες της μετανάστευσης καθώς και τις πολιτικές ένταξης. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των παραδοσιακών πολιτικών. Με τις περικοπές της πολιτικής συνοχής και την ε, πολιτική, τη γεωργική, που είναι η καρδιά της Ευρώπης. Προσοχή. Ε, ούτως ή άλλως, οι εθνικές συνεισφορές δεν μπορούν να αυξηθούν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει το θάρρος να χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους βάζοντας για πρώτη φορά ένα πραγματικό carbon tax και μια ένα πραγματικό και θαραλέο web tax, ψηφιακό φόρο. Ευχαριστώ τον κύριο Πεντιτσίνη. Ακούσαμε τις πολιτικές ομάδες και τώρα ο κύριος Όλμπριχτ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν είναι ποτέ καθαρά δημοσιονομική. Μιλάμε θέματα που αφορούν τις μελλοντικές μας πολιτικές και τώρα είμαστε σε περίοδο μετά τον Brexit. Πολλοί λένε τώρα ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα, να αναθεωρήσουμε κάποια άλλα. Αλλά ο τρόπος βελτίωσης είναι διαφορετικός κάθε φορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι μετά το Brexit η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει το επίπεδο δραστηριοτήτων της και φιλοδοξιών της ε, ακόμα και να τις επεκτείνει. Δηλαδή αυτό που κάναμε και αυτό που χρειάζεται για το μέλλον. Στο Συμβούλιο το βλέπουν διαφορετικά. Κάποιοι λένε ότι θέλουν μικρότερο προϋπολογισμό και άλλες λένε ότι θέλουν λιγότερες δραστηριότητες σε επίπεδο ένωσης. Θέλουν μικρότερο εύρος δραστηριοτήτων. Θέλουν να ξαναγυρίσουν στην παλιά βρετανική ιδέα, δηλαδή επανεθνικοποίηση κάποιων πολιτικών. Γι' αυτό δεν θέλουν να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα. Δεν πρόκειται μόνο για τον προϋπολογισμό, αλλά και για την Ένωση μετά τον Brexit. Θέλουν να είναι μικρότεροι ως προς το εύρος της. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά πλειοψηφία, δεν συμφωνεί με τη στάση αυτή. Μετά τον Brexit η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραιτηθεί από το επίπεδο των φιλοδοξιών της, γιατί αυτό θα αποδείκνυε ότι δεν μπορούμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις. Πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τις πρόσθετες αλλαγές και τις πρόσθετες προκλήσεις ε, μέσα από τους ίδιους πόρους. Εμείς στο Κοινοβούλιο δεν θα συμφωνήσουμε με δράσεις που μικραίνουν και κάνουν πιο αναποτελεσματική την Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για δυόμιση λεπτά η κυρία Μάρκες. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, πρόσωποι του Συμβουλίου. Τώρα, Σημαντικό είναι να ε, συγκεράσουμε προτεραιότητες με δαπάνες. Θα πρέπει να βρεθούν πολιτικοί συμβιβασμοί ε, που θα αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας υπέρ των πολιτών. Πρέπει να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Και αυτή η χρονική περίοδος ε, συμπεριλαμβάνει τεράστιες προκλήσεις. Πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ε, μια άσκηση κατά την οποία κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να βγει από τη βολή του και από τους εθνικούς εγωισμούς του. Γίνεται αυτό. Το είδαμε στη μακρά ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές ε, μπόρεσαν να συγκεραστούν τα εθνικά με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Υπάρχουν για μας πολιτικές προτεραιότητες και πρέπει αυτές να συνεχίζονται. Ε, δεν είναι κενά λόγια αυτά. Αυτά είναι η απήχηση πολιτικής βούλησης. Παραδείγματα συγκεκριμένα. Θέλουμε επενδύσεις για την οικονομική ανάπτυξη, για περισσότερη απασχόληση. Έχουμε το InvestEU, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες, έχουμε το πρόγραμμα συνοχής, θέλουμε να περάσουμε στην ψηφιακή αλλαγή, έχουμε το Digital Europe, Έχουμε συνεργασία των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών μας. Θέλουμε να βελτιώσουμε την κινητικότητα των νέων. Βλέπε Εράσμους. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ε, το μηχανισμό Just Transition. Και ο κατάλογος ε, μπορεί να συνεχιστεί επί μακρόν. Για όλα αυτά χρειάζονται λεφτά. Αυτά που έχουμε να διαθέσουμε δεν επαρκούν. Θα πρέπει να αυξήσουμε τα κονδύλια. Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες της Ένωσης ε, πρέπει να καλύπτονται και χρειάζονται ήδη οι πόροι που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε θεσμική κρίση, αλλά δεν θα εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που δεν ανταποκρίνεται στις πολιτικές μας προτεραιότητες και δεν επιτυγχάνει συμφωνία επί των ιδίων πόρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χαγέρη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, κύριε Υπουργέ. Μετά από δύο χρόνια ε, αναβολ... καθυστέρησης αντιμετωπίζουμε αυτό το... Ε, βρισκόμαστε σε μια καμπή της ιστορίας μας. Το... Οι συλλογικές προκλήσεις είναι γιγαντιές. Απαιτούν ε, ταχείες ε, προσπάθειες, χωρίς κοινό μέτρο, όλοι το γνωρίζουμε. Ωστόσο, μετά από πάνω από 70 χρόνια συμβίωσης, το 1% δεν τίθεται ένα αμφιβόλο. όλοι διαρωτώνται πόσα τα κράτη πόσα πρέπει να δώσουν και πόσα θα πάρουν. 0,02% ε, εδώ, εκατό εκεί. Για ορισμένες χώρες το ζούμενο είναι η μείωση της εθνικής εισφοράς και αυτό ενθαρρύνεται και από το ίδιο μας το σύστημα της χρηματοδότησης. Το 80% των εθνικών εισφορών, αυτό το σύστημα παρούσας χρηματοδότησης είναι διαστραμμένο. και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι μεν και οι δε, ε, δημιουργούνται ακόμα πιο ε, πολύπλοκα συστήματα. Το έργο του Πρόεδρου του Συμβουλίου δεν είναι απλό, αλλά έχει όλη μα την υποστήριξη, όπω και η Επιτροπή. Προκειμένου να πετύχουμε τον τεραγωνισμό του κύκλου, θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη των ιδίων πόρων. Με του ιδίου πόρου που κάποτε ήταν η ευρωπαϊκή ταυτότητα, με τον τρόπο αυτό οι εθνικέ εισφορέ θα μειωθούν. Άρα θα βρούμε όλοι κερδισμένη, όπω είπε η κυρία Πρόεδρο, Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχυθεί με μεγαλύτερη ε, αυτονομία οικονομική, προκειμένου να καλύψει προτεραιότητές της. Ε, είναι σημαντική, είναι κρίσιμη συγκυρία το σύστημα τη χρηματοδότησή μα διανύει μια επαξιακή κρίση. Ας είμαστε ξεκάθαροι, χωρί μεταρρυθμίσει. Ε, έχουμε τον κίνδυνο να αποτύχουν όλες μας, να όλε όλες μας οι ελπίδες. Η συνάντηση κορυφής Φεβρουαρίου θα είναι κρίσιμη προκειμένου να προσμετρήσουμε την ε, πραγματική υπόσταση των φιλοδοξιών των κρατών ε, έναντι του Κοινοβουλίου. Και εγώ δεσμεύομαι να υπερασπιστώ αυτέ τι μεταρρυθμίσει για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά, ο κύριος Μπέι. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι η μετάφραση των δικών μας πολιτικών προτεραιοτήτων. 1,1% ή 1,3% του ΑΕΠ, 1.200 ε, δις ε, ευρώ κλπ. Ε, το Brexit, τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ δημιουργούν ένα έλλειμμα. Ε, τι θα κάνουν, τι θα σκεφτούν οι πολίτες μας και ο υπόλοιπο κόσμος ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία εγκατέλειψε η Μεγάλη Βρετανία ε, και η οποία πρόκειται να φορτωθεί μελλοντικά την Αλβανία και τη Βόρεια ε, Μακεδονία. Ε, λιγότερο το 1% αφιερώνεται στην προστασία των συνόρων. Σήμερα το πολιτές και οι στόχοι της Επιτροπής ε, αφορούν την θυσία τελικά της γεωργίας μας και 33% το προπολογισμό για τις κλιματικές αλλαγές. 300 δις ε, ευρώ για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων η οποία υποσκάπτεται από τις ελεύθερες αλλαγές ε, σε διεθνή κλίμακα. Κυρία Φοντερ μας λέτε ότι θέλετε να δημιουργήσετε καταρχήν αυτόν τον προπολογισμό μαζί με τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά θα πρέπει να τους ακούσετε. Αυτοί θέλουν οικονομική κατοχήρωση των έλεγχων των συνόρων. Δεν θέλουν ιδίους πόρους, ε, ένα ευρωπαϊκό φόρο ε, που επιβαρύνει χώρες όπως η Γαλλία που το 45% ε, του ΑΕΠ είναι αντιστοιχεί σε υποχρεωτική φορολόγηση. Δεν πρέπει με τον τρόπο αυτό να συγκαλύπτουμε την ανυμπόρια μας. Δύο λεπτά, ο κύριος Ευχαριστώ. Τώρα θα πρέπει να δοθούν μάχες ε, ε, από τα κράτη-μέλη και τη Γερμανία και την κυρία Μέρκελ. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κρύβονται ε, πίσω από μειώσεις υπονομεύοντας το μέλλον της Ευρώπης ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, την ανεργία των νέων, θέλουμε να επενδύσουμε στην ψηφιοποίηση και την έρευνα. Οι πράσινοι θέλουν. Γι' αυτό θα κρίνουμε την πρόταση που θα υποβληθεί με βάση αυτά, γιατί το 1,0% ή 1,07% είναι λίγο, σημαίνει περικοπές. Εμείς χρειαζόμαστε κοινέ επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, να δώσουμε περισσότερα, περισσότερα δίκαια τα, τα ε, κονδύλια, λιγότερο για τον άνθρακα, περισσότερο ε, για το αέριο και ανανεώσιμες πηγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να προωθεί τη δημοκρατία και τις αξίες. Όταν ε, καταπατώνται όλα αυτά, δεν καλύπτονται με τα κονδύλια. Ε, ε, δεν θα, δεν ε, εγκρίνει το Κοινοβούλιο έναν προϋπολογισμό έμπνευσης Όρμπαν. Εμείς βλέπουμε με επιφυλακτικότητα της, τη γερμανική πρόταση και τη γερμανική πολιτική σήμερα που στηρίζεται στις εξαγωγές και ωφελείται από τις επενδύσεις όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Θέλουμε η γερμανική κυβέρνηση να ταχθεί υπέρ ενός ε, στιβαρού ε, νοσιακού προϋπολογισμού ε, ε, έτσι θα δείξει ότι επενδύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να δοθούν 20 ή 30 cents παραπάνω ε, οι πολίτες ούτως ώστε να έχει έναν στιβαρό προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανόβερφελτ, 1,5 λεπτό. Κύριε, κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. μας δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία ε, μετά την επανεκλογή του νέου κοινοβουλίου κατά 60% νέα μέλη, η Κομισιόν με νέες φιλοδοξίες και οι αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι ε, σπάνιο να βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Να πω επίσης ότι αυτό το κοινοβούλιο με 60% νέα μέλη ε, μπορεί να συμπαρασταθεί στους φιλόδοξους στόχους της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν από την κυρία Φόντερ Λάιεν. Ε, παρουσίασε σημαντικές προτεραιότητες για ένα μέλλον ανταγωνιστικότητας και ευημερία. Οι φιλοδοξίες αυτές απαιτούν χρήματα, γι' αυτό χρειάζεται σωστός προϋπολογισμός. Ακούγοντας κάποιους επιτρόπους ε, να σχολιάζουν, να μιλούν για αυτό το θέμα, λένε ότι πρέπει να προωθηθεί η πράσινη συμφωνία με λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι ανεύθυνο. Τέτοιου είδους δηλώσεις νομίζω ότι θα τρομάξουν ε, τους ε, πιθανούς επενδυτές. Παράλληλα, η Ευρώπη πρέπει να φροντίσει ότι θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότητα κάθε προγράμματος. Θα πρέπει κάθε ευρώ που δαπανάτε να προσφέρει προσθέμενη αξία στους πολίτες. Ο Μαρζή, 1,5 λεπτό. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ότι δεν έχετε καμία ιστορική αίσθηση εσείς οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Έχουμε μεγάλες ε, Δημογραφικέ, οικονομικέ και κλιματικέ αλλαγέ στον κόσμο. Και αυτό υποχρεώνει την Ευρώπη να κάνει ένα άλμα προ τα εμπρό. Υπάρχουν όλο και περισσότεροι πειρασμοί για αναδίπλωση. Και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουμε αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων που δεν είναι στο ύψο αυτή τη ιστορική στιγμή και που συμπεριφέρονται σαν μικροί διαχειριστέ ενό μικρού συνεταιρισμού. Δεν υπάρχουν οι μεγάλε φωνέ, δεν υπάρχει το κουράγιο για να ανοίξουμε το δρόμο για μια Ευρώπη που θα έχει ξεφορτωθεί τη λιτότητα, που θα είναι ικανή να διδαχθεί από τις πιο σημαντικές υποσχέσεις ε, αυτού του αιώνα και να προχωρήσει. Αντί να προχωρήσει όμως, υποχωρεί. Με ένα μικρό προϋπολογισμό η Ευρώπη θα υπαναχωρήσει τα επόμενα δέκα χρόνια με τι περικοπέ στον προπολογισμό τη κοινή γεωργική πολιτική και στην πολιτική συνοχή. αυτό τι σημαίνει. Ότι θα έχουμε λιγότερη συνοχή, άρα λιγότερη ανάπτυξη, λιγότερες επενδύσεις, λιγότερες θέσει απασχόλησης, περισσότερες ρογμέ, περισσότερα προβλήματα. Η πολιτική συνοχή είναι η πολιτική του μέλλοντο. Για τον προπολογισμό του 2014-2020, περίπου 100 δις ευρώ επενδύθηκαν στο περιβάλλον και στο κλίμα χάρη σε αυτή την πολιτική, μέσω αυτή της πολιτικής. Ευχαριστώ. Κύριο Μαρζέ, υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Από τον κύριο Μάρκες. Τη δέχεστε? Παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα στον κύριο Μάρκες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Όμορζε, στην Πορτογαλία, την πατρίδα μου, εμείς γυρίσαμε τη σελίδα της λιτότητας, φέραμε ελπίδα στη χώρα και σε πολλούς Ευρωπαίους που είδαν ότι είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε τη λιτότητα. Στο νέο αυτό προϋπολογισμό πρέπει να υπάρχει μια νέα ελπίδα για την Ευρώπη θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ε, υποσχέσεις που δώσαμε. Να έχουμε πιο φιλόδοξη Ευρώπη. Και ο εξυγχρονισμός είναι σημαντικός των πολιτικών ε, στις οποίες πιστεύουμε. Ευχαριστώ. Διακόπτη ο Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι ήταν σαφής η ερώτηση. Κύριε Ομέρτζε, θέλετε να απαντήσετε. Συνάδελφε, Πέδρο Μάρκες, νομίζω ότι τα οράματά μας συμπίπτουν. η πολιτική συνοχής όντω είναι μια πολιτική που θα συμμετάσχει στις νέες προτεραιότητες που καθορίζονται σήμερα. Αυτή η διάκριση ανάμεσα σε παραδοσιακές και νέες πολιτικές είναι μια διάκριση που δεν έχει πραγματικά θεμέλια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδάκης, ένα λεπτό η συζήτηση του προπολογισμού είναι σημαδεμένη από μεγάλα συμφέροντα ναρκοθετημένη για το λαό. εντείνεται με ταμεία και μηχανισμούς η στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής ένωσης διαγωνίζονται ποιες χώρες κλάδοι και όμιλοι θα ωφεληθούν περισσότερο από τους ανταγωνιστές τους στο έδαφος του brexit. επιδοτούνται οι όμιλοι στο όνομα της ψηφιακής μετάβασης για να διευρυνθούν η εργασιακή γαλέρα οι απολύσεις και η φτώχεια με δούριο ύπο τα κονδύλια της ευρωπαϊκής ένωσης στην ελλάδα η κυβέρνηση της νέας δημοκρατίας σε συνέχεια του σύριζα κλείνει τις λιγνητικές μονάδες οδηγώντας στην ανεργία πάνω από πέντε χιλιάδες εργάτες στερώντας από τη χώρα τη δυνατότητα αξιοποίησης εγχώριων πηγών ενώ ενισχύεται η εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια που ακριβοπληρώνει ο λαός. με όχημα το green deal και τη νέα ακόμα πιο αντιδραστική ΚΑΠ, προωθείται η κερδοφορία των ομίλων και το ξεκλήρισμα των βιοπαραστών αγροτών με μείωση των ενισχύσεών του. δεν μας ξαφνιάζει ο ταξικός αντιλαϊκό χαρακτήρας του προπολογισμού. γι' αυτό στηρίζουμε την πάλη των εργαζομένων για τις δικέ του ανάγκες ενάντια σε επιχειρηματικού ομίλους και αντιλαϊκή πολιτική. Η κυρία Γραπίνη θέλει να υποβάλει μια ερώτηση. Δέχεστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ συνάδελφοι, είσαστε αντίθετο στην κοινή γεωργική πολιτική. Μας λέτε ότι κάποιοι αποφελούνται από αυτό. Αλλά με το νέο προπολογισμό, με το νέο ε, πουδουπού θα πρέπει να μειωθεί και αυτός ο προπολογισμό, δηλαδή. Θα πρέπει να βρούμε ε, τους πόρους όμως από τη φοροδιαφυγή π.χ. για να μην μειώσουμε το προβληματισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Ο κ. Παπαδάκης θέλει να απαντήσει. Κάθε περίπτωση η ωφελημένη και της νέας ΚΑΠ θα είναι επιχειρηματική όμιλη άλλωστε ο πυλώνας των επενδύσεων των καπιταλιστικών επενδύσεων είναι αυτός που ενισχύεται και αυτό που συρρυκνώνεται είναι το ποσοστό των ενισχύσεων της μικρομεσαίας αγροτιάς. αυτοί είναι τα θύματα για άλλη μια φορά και οι όμιλοι είναι αυτοί που κερδίζουν και αυτή είναι η νέα γραμμή που συνεχίζει και τις προηγούμενες καπ και θα εντείνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα για τους μικρομεσαίους αγρότες που ο μόνος δρόμος τους είναι να οργανώσουν την πάλη τους πριν να είναι αργά. Ο κύριος Φερνάντες, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς περιμένουμε από τον Νοέμβριο του 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τέλος πάντων, κάλλια αργά παρά ποτέ. Χρειαζόμαστε επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για συνεκτική, ανταγωνιστική, παραγωγική Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται για βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και παράλληλα πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Χρειάζονται νέοι ίδιοι πόροι. Αυτό είναι η λύση. Για να ε, σταματήσουν οι συντηρητικές λογικές. Αυτό χρειάζεται. Όμως όχι σε βάρος του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η αρχή μας είναι απλή. Όποιος δεν πληρώνει πρέπει να καθίσταται υπόλογος. Χρειαζόμαστε ε, φόρο ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ε, φόρο για ψηφιακές επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε επίσης